Pan Przewodniczący! Wznawiam posiedzenie. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίασή μα. Τα πρακτικά τη χθεσινή συνεδρίαση είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν σχόλια. Δεν βλέπω κανένα να θέλει να σχολιάσει, οπότε εγκρίνω τα πρακτικά. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια μας διάταξη είναι η δήλωση του Ευρωπαϊκού